Okay. Good afternoon everybody. Καλό απόγευμα σε όλους. Ζητώ συγγνώμη που έχουμε καθυστερήσει. Θα μπορούσαμε να είχαμε ξεκινήσει νωρίτερα. Εάν είχα καταλάβει ότι έχουμε χωρίσει τη συνεδρία σε δύο κομμάτια, ένα από τις 3 έως τις 3.30 και το άλλο από τις 3.30 μέχρι τις 6.30. Ε, ξεκινούμε λοιπόν τη συνεδρίαση, τη συνεδρίαση της Επιτροπής ΦΑΜ και θα έχουν μετά την ε, κοινή δημόσια κρόση μαζί με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Ο κύριος Αγγιλάρ, πρόεδρος της ΛΥΜΠΕ, θα καταφτάσει πολύ σύντομα. Θα ξεκινήσουμε όμως με το σημείο 12 της ημερήσιας ε, διάταξης ε,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 έχει τη δυνατότητα να δει τι δουλειά έχουν κάνει τα κράτη-μέλη. Ε, αφότου η Ουγγρική Προεδρία ξεκίνησε το πλαίσιο ε, για, ε, την, για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρωμά που αφορά τα 40 εκατομμύρια των φτωχότερων ανθρώπων της Ευρώπης που είναι καταγωγής Ρωμά. Πολλά από αυτά τα αστικά γκέτο και ε, στις πόλεις αλλά και στην Υπεθρό βλέπουμε ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί στους, ε, ε, στα μέρη αυτά. Πολύ λίγη πρόοδος έχει σημειωθεί και γι' αυτό το Κοινοβούλιο δεσμεύεται να συνεχίσει να βοηθάει την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν αποτελεσματικά το σχέδιο δράσης και να μην ακούμε μόνο λόγια, ιδέες και να σπαταλάμε χρήματα. Κάτι που είδαμε την τελευταία 20 με πολύ ισχυρά αποτελέσματα. Αυτή λοιπόν η πρώτη εξέταση των ε, εθνικών ε, στρατηγικών και βέβαια μιλάμε για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, διότι όταν μιλάμε για την ε, μείωση της ε, δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα να λύσουμε το πρόβλημα μέσα σε λίγα χρόνια. Ε, ωστόσο, πιστεύουμε ότι η πρόοδος ε, δεν είναι πολύ μεγάλη, γιατί προσπάθησα να εξετάσω τη διάσταση του φύλου στην έκθεσή μου, διότι εάν εξετάσουμε τη, τους πιο ευάλωτους ανθρώπους από αυτά τα 40 εκατομμύρια, τις γυναίκες και τα παιδιά και τους μη Ρωμά που ζουν σε, αυτές, σε αυτά τα γκέτο, θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε στα κράτη-μέλη μια συνολική εικόνα. Ποιες πολιτικές έχουν σχεδιαστεί σωστά, έχουν χρηματοδοτηθεί επαρκώς, ε, έχουν παρακολουθηθεί σωστά, έχουν σχεδιαστεί σωστά και όπου υπάρχει συμμετοχή και των Ρωμά. Αυτά λοιπόν είναι τα ερωτήματα που θέσαμε και ζητήσαμε από διάφορες οργανώσεις ε, να κάνουν έρευνες. Ε, και επιτρέψτε μου να πω ότι βρήκαμε την ε, συνεισφορά αυτών των οργανώσεων πολύ χρήσιμη στο πρώτο μέρος του εγγράφου μιλάμε γενικά, στο δεύτερο μέρος ε, μιλάμε ιδιαίτερα για τις ε, γυναίκες και γι' αυτό χρειαστήκαμε τα ε, αναλυτικά στοιχεία της ΕΦΕΡΑ. Και διαπιστώσαμε ότι ο κίνδυνος φτώχειας για οικογένειες Ρωμά με πάνω από τέσσερα παιδιά είναι πολύ μεγάλος. Διαπιστώσαμε όμως ότι, ε, ότι στις μονογονεϊκές οικογένειες ήταν πολύ μεγαλύτερος ο κίνδυνος αυτός ε, και επίσης ότι οι ηλικιωμένε ε, ανήπαντρες ε, Ρωμά είναι από τις πιο ευάλωτες κατηγορίες και επίσης οι περισσότεροι άνεργοι Ρωμά είναι γυναίκες. Επίσης είδαμε πολύ περισσότερο αναλφαβητισμό Είδαμε πολλές ε, εγκυμοσύνες ε, κατά την εφηβεία ή μη σχεδιασμένε, μη προγραμματισμένες ε, εγκυμοσύνες στις γυναίκε αυτές. Και επειδή θέλουμε να καταπολεμήσουμε την ε, φτώχεια βλέπουμε ότι ο αυξημένος ε, κίνδυνος ε, εμπορίας ανθρώπων, η πορνεία κτλ. αποτελούν επίσης μέρος της έκθεσής μας. Όσον αφορά την, τη συμπερίληψη της διάστασης του φύλου και την παρακολούθηση των θεμάτων αυτών, την, ε, χρειαζόμαστε πολύ πιο στοχευμένες δράσεις όσον αφορά την ε, μείωση της ε, της στα παιδιά. πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το θέμα των έφηβων μητέρων, των κοριτσιών που, νωρίς, που εγκαταλείπουν νωρίς στο σχολείο και πρέπει να ε, εξετάσουμε και την ε, ένταξη στην αγορά εργασίας. Ε, τα εργοστάσια, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θέλουν να προσλάβουν τις γυναίκες αυτές. Η διαβίω εκμάθηση λείπει τελείως από τις περιοχές αυτές και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα και βλέπουμε έμεσες και άμεσες διακρίσεις εις βάρος των γυναικών αυτών. Θα πρέπει να συζητηθούν τα θέματα αυτά ώστε η Κομισιόν να καταλάβει τι μήνυμα πρέπει να στείλουμε στα κράτη-μέλη. Και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την Edit Power για τη γνωμοδότησή της. Διότι η γνωμοδότηση αυτή εξηγεί ποια είναι τα βασικά προβλήματα, η εκπαίδευση και η δουλειά και η απασχόληση η πρόσβαση σε θέσεις απασχόλησης όταν εγκαταλείπει κανείς ε, την ε, διευρυμένη οικογένειά του. Και θα κλείσω εδώ να σας ευχαριστήσω για όλες τις συνεισφορές που έχω λάβει μέχρι στιγμής από τους συναδέρφους και από ε, μη κυβερνητικές οργανώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε το λόγο ε, στους Κυρία Κλεβέτη, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όσον αφορά την έκθεση αυτή, θα συνεισφέρω και εγώ ως σκιώδης εισηγήτρια για τους ε, σοσιαλιστές. Όπως και η εισηγήτρια και εγώ θεωρώ το θέμα αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έχει άμεση ανάμειξη στον εντοπισμό λύσεων για την ένταξη των Ρωμά είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Η απόφαση αυτή έχει επιτρέψει στα κράτη-μέλη να συντάξουν αυτές ε, τις ε, εκθέσεις αναχώρα για το θέμα αυτό και έχοντας διαβάσει τις εκθέσεις αυτές μπορώ να πω ότι υπάρχει μικρή αναφορά στα ζητήματα του φίλου. Ωστόσο, μπόρεσα να εντοπίσω ορισμένες βέλτιστες πρακτικές σε συγκεκριμένες χώρες και θα τις κατονομάσω, διότι δεν θέλω να τις ξεχάσω. Εκτός από αυτά που ήδη αναφέρθηκαν από τη συνάδελφό μου, πιστεύω πως είναι επίσης σημαντικό να ασχοληθούμε με τους τέσσερις κύριους προβληματικούς τομείς. Την απασχόληση, την εκπαίδευση, την υγεία και τη στέγαση των γυναικών Ρωμά. Υπάρχουν επίσης δύο πολύ σημαντικά θέματα. Η ελεύθερη μετακίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η καταπολέμηση των στερεοτύπων για, την, ε, για τους ε, Ρωμά γενικότερα. Όλοι πρέπει να συνεισφέρουμε και να βοηθήσουμε για να αναλυθούν αυτά τα εκκρεμή ζητήματα καλόπιστα και να βρεθεί μια ευρωπαϊκή λύση. Ως εκπρόσωπος ε, της Ρουμανίας, ενός ε, κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μεγάλη κοινότητα Ρωμά, μπορώ να συνεισφέρω με την εμπειρία από τη Ρουμανία. Εμείς έχουμε μια μεγάλη ιστορία συνύπαρξης με την κοινότητα των Ρωμά και αυτό έχει βοηθήσει τους Ρουμάνους να μάθουν και τις καλές και τις άσχημες πλευρές της κοινότητας αυτής. Δεν πρέπει να ασκούμε κριτική ανεξαρτήτως σε όλους τους Ρωμά, πρέπει να ξέρουμε τις ε, λεπτομέρειες, διότι είναι μια ιδιαίτερη κοινότητα με τις δικές της ιδιαιτερότητες και χρειάζεται να βρούμε ευρωπαϊκές λύσεις για τα προβλήματά τους. Θα σταματήσω όμως εδώ, διότι θα υποβάλω τροπολογίες για την έκθεση αυτή και θα συνεργαστώ με τους συναδέλφους μου για την ολοκλήρωση της έκθεσης. ενδιαφέρομαι για την έβρεση λύση στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μπάουερ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κάποιες ε, σύντομες ε, παρατηρήσεις. Σήμερα στην Επιτροπή Απασχόλησης συζητήσαμε τη γνωμοδότηση για την έκθεση αυτή. όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Απασχόλησης, το θέμα της δουλειάς δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι είναι απαραίτητο να κάνουμε σαφή διάκριση ανάμεσα στην απασχολησιμότητα, την πρόσβαση στη, σε θέσεις απασχόλησης, ε, και τις διακρίσεις. Τα φαινόμενα αυτά συνδέονται μεταξύ τους, αλλά είναι σαφές να πούμε τι είναι η απασχολησιμότητα, έχοντας κατά νου το τεράστιο ποσοστό αναλφαβητισμού μεταξύ των γυναικών Ρωμά και το χαμηλό ποσοστό απασχόλησης. Μόλις το 24% έχουν δουλειά από τις γυναίκες Ρώμα. Πρόκειται λοιπόν ε, για μια ειδική περίπτωση στην αγορά εργασίας και αποτελεί μεγάλη πρόκληση. Θα πρέπει καταρχήν να εξετάσουμε το θέμα της απασχολησιμότητας διότι για, ε, το, για, μεγάλο, για μεγάλες ομάδες ανειδίκευτων ανθρώπων δεν θα έχουμε δουλειά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς λοιπόν μπορούμε να αναβαθμίσουμε ε, τα προσόντα των Ρωμά. Και υπάρχει το θέμα της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Υπάρχει. Και το θέμα να δημιουργήσουμε στα κοινωνικά συστήματα κίνητρα για εργασία. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις μεγάλες οικογένειες και τις ε, ανήπαντρες μητέρες. Διότι η οικονομική ανεξαρτησία ε, ε, είναι πολύ χαμηλή μεταξύ των γυναικών Ρωμά. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε σαφώς ότι αυτοί οι στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί και είναι πολύ σημαντικές αυτές οι προκλήσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στην εκπρόσωπο της ε, Κομισιόν, την κυρία Παπαμιχαλοπούλου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Παπα Μιχαλοπούλου με λένε. Λίνα όμως είναι πιο εύκολο. Καταρχάς να πω ότι η Επιτροπή καλωσορίζει την πρωτοβουλία της Λίβια για την έκθεση αυτή. Σίγουρα η Επιτροπή έχει σαφή επίγνωση ότι οι γυναίκες Ρωμά είναι ιδιαίτερα τροτές τόσο στη σχέση άνδρα-γυναίκας, όσο και στη σχέση Ρωμά ευρύτερης κοινωνίας. Δεν θα ήθελα να παραπέμψω στα στατιστικά που έχουμε σε λεπτομέρειες, διότι προέρχονται από την πρόσφατη έρευνα της ΦΡΑ και ξέρω ότι αργότερα στην ακρόαση θα μιλήσει η ΦΡΑ και θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα αυτά. Θα περιοριστώ λοιπόν στο να πω ότι εντοπίσαμε πως ε, υπάρχει ένα σοβαρό το ζήτημα στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην υγεία. Οι γυναίκες υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις. Θέσαμε το θέμα αυτό στην έκθεσή μας. Ταυτόχρονα πρέπει να αποδεχθώ ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο θέτει, αντιμετωπίζει το θέμα αυτό μόνο περιστασιακά, δεν αντιμετωπίζουμε πραγματικά το έμφυλο ζήτημα. Στην έκθεση του Ιουνίου, ωστόσο, πα, παρακινήσαμε τα κράτη να, υπάρξει, να κάνουν δουλειά στον τομέα αυτό, ιδιαίτερα στον τομέα των πολλαπλών διακρίσεων. Στην πρόταση που πρόσφατα υποβάλαμε στο Συμβούλιο ω σύσταση, περιλάβαμε ένα τμήμα, το 3-5, ειδικά για το θέμα της προστασίας των γυναικών και των παιδιών Ρωμά συμπεραίνω ότι περιμένουμε, κλείνω περιμένοντας την τελική έκφραση και θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Γιαρόκα που ήταν πολύ καλή φίλη στην μονάδα συντονισμού των Ρωμάτων τα τελευταία χρόνια. Eh, Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στην κυρία Γιαρόκα εάν θέλει να ε, κάνει κάποιες ε, τελικές παρατηρήσεις. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Δεν θα μακρηγορήσω. Απλά να πω ότι εμείς θέλαμε να δούμε τα φτωχότερα και πιο περιθωριοποιημένα στρώματα των φτωχότερων της Ευρώπης. Γι' αυτό είδαμε τις γυναίκες και την έμφυλη διάσταση. Το κάναμε όμως και γιατί αυτό είναι κάτι που λείπει σε όλες τις εθνικές ε, στρατηγικές και αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό γιατί ξέρουμε τα ευρήματα των ερευνών. Οι γυναίκες στην περίοδο κρίσης για πολλές κοινότητες ζωμά αποτελούν τη μόνη διέξοδο ε, με τον υπόλοιπο κόσμο. Η ΦΡΑ στην έκθεσή της έδωσε κάποια νέα στοιχεία. Μαθαίνουμε, για παράδειγμα, ότι σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην υγεία, περισσότερο πλήττονται οι άνδρες Ρωμά παρά οι γυναίκες. Αυτά μας λέει η ΦΡΑ. Ο στόχος μας λοιπόν πρέπει να είναι να σταματήσουμε αυτό το φαύλο κύκλο φτώχειας, περιθωριοποίησης, κληρονομιάς της φτώχειας. Το μήνυμα που πρέπει να περάσει από εδώ είναι ότι η μία αγνώριση του γεγονότος ότι οι γυναίκες Ρωμά μεγαλώνουν τα παιδιά τους χωρίς να έχουν στα περισσότερα κράτη-μέλη τουλάχιστον κάποιο εισόδημα για το σκοπό αυτό, δημιουργεί μία διάκριση που δυσχεραίνει τη δυνατότητα των γυναικών Ρωμά να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους, το ρόλο, να παίξουν το ρόλο τους. Να δείξουμε λοιπόν στα κράτη-μέλη ότι έχουν την ευθύνη και την ανάπτυξη αυτών των παιδιών Γι' αυτό θεωρούμε πολύ σημαντικά να δώσουμε έμφαση στις γυναίκες Ρωμά και τα παιδιά Ρωμά στην έκθεσή μας, δείχνοντας και τις άλλες δυσκολίες που υπάρχουν, παρότι υπάρχουν και εθνικά προγράμματα για Ρωμά και κάποια λεφτά για τα προγράμματα αυτά. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Η Επιτροπή Γυναικών είναι πολύ τυχερή που έχει τόσο καλή εισηγήτρια για τόσο σημαντικό θέμα. Καλή τύχη στη δουλειά σας. Κύριε Γιάλογα και ευχαριστούμε. I will now read out the Uh, διαβάσω τις προθεσμίες τώρα για την υποβολή των τροπολογιών. 24 Σεπτεμβρίου 12 το μεσημέρι. Η Επιτροπή Γυναικών θα ψηφίσει την έκθεση αυτή στις 14 Οκτωβρίου. Στην Ολομέλεια μάλλον του Νοεμβρίου, αλλά παίζει ακόμα. Αφήνουμε το σημείο αυτό. Κάνουμε ένα διάλειμμα δύο λεπτών πριν ξεκινήσει η κοινή ακρόαση.